Τη δήλωση αυτή την κάνω εξ ονόματος της συναδέλφου μου Χρισταλίνας Γεωργίευα που είναι υπεύθυνη για ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση των θεομηνιών. Είναι φανερό το γιατί χρειάστηκε η αντικατάσταση, γιατί η Επίτροπος Γεώργιεβα είναι στη Χιλή από χθε για να επισκεφθεί τις περιφέρειες που έχουν πληγεί και να δει πώς εργάζονται εκεί οι διάφοροι ανθρωπιστικοί εμπειρογνώμονες. Μόλις έφτασε στο Σαντιάγο έσπευσε στον τομέα του τσουναμίου και στην Κονσεψιόν. Κατά την επίσκεψή της συνάντησε εκπροσώπους Μίκη όμικρον που εργάζονται εκεί και με τις αρχές της Χιλής που είναι παρούσες εκεί. Η Επίτροπος Γεωργίευα θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο Μπαρόσο και στην ενθρόνηση του Προέδρου. Ο σεισμός και μετά το τσουνάμι που έπληξαν τη Χιλή το πρωί του Σαββάτου είναι μια τρομερή τραγωδία. Οι τελευταίοι επίσημοι αριθμοί λένε ότι τουλάχιστον 520 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αναμένεται να αυξηθούν οι αριθμοί. Πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν πληγεί. Η ζημία στις υποδομές είναι τεράστια και 500.000 σπίτια επίσης έχουν καταστραφεί. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Χιλή, Μαριάνο Φερνάντες, δέχτηκε την ίδια μέρα ήδη τα συλληπιτήριά μα. Μόλις ακούστηκαν τα νέα για το σεισμό, κινητοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης. σε όλες τις χώρες που αφορούσε και το MIC ήδη αμέσως είχε νέα που διέδωσε και ταύτισε στόχους που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν. Η Επίτροπος Γεωργίευα πήγε στην αίθουσα κρίσεων αμέσως για να δει πώς θα διαχειριστεί την κρίση αυτή. Πολλές χώρες μέλη έκαναν προτάσεις βοηθείας χορήγησης προσωπικού, υλικού, η Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες χώρες, Φιλανδία και υλικά όπως γεννήτριες, κουζίνες ε, κλπ. από την Αυστρία και άλλες χώρες. Οι αρχές της Χιλής δήλωσαν ότι δέχονται τις προσφορές αυτές και το σύστημα άμεσης και ανθρωπιστικής βοηθείας της Ένωσης κινητοποίησε μέσω το γραφείο στη Μανάγουα για να χορηγηθεί άμεση ανακουφιστική βοήθεια που να χορηγηθεί στην περιοχή του σεισμού. Ήδη από την Κυριακή το πρωί ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές και συμφωνίες για δωρεές, ανθρωπιστικές δωρεές έχουν ήδη συναυθεί. Το Telecom San Frontier από τη Γαλλία δέχτηκε όπως και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός να χορηγήσει τηλεπικοινωνιακά υλικά και ιατρική βοήθεια. και από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου έφτασαν εμπειρογνώμονές μας στη Χιλή για να συναντήσουν τις αρχές και να δουν ποιες είναι οι ανάγκες. Και την επόμενη μέρα, τρίτη δηλαδή, προσθέθηκαν και άλλοι δύο και ύστερα και άλλοι. Μία ομάδα έξι εμπειρογνωμόνων επίσης έχει σταλεί, τέσσερις από τους οποίους είναι ήδη στη ζώνη του σεισμού στην Κονσεψιόν και άλλοι στο Σαντιάγο συνεννοούνται με τις αρχές και συντονίζουν τις προσπάθειες της Ένωσης με εκείνους. Γίνονται αξιολογήσεις με ορισμένες ε, με όλα τα αρμόδια όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Και τώρα η κυρία Στρίφλερ από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί, όπω ελέγχθη, ο σεισμό ε, στην Χιλή, του οποίου ένταση ήταν υψηλότερο από εκείνον που έπληξε την ΑΕΤ και που η Χιλή επιλύγηκε από ένα τσουνάμι, είχε αποτελέσματα λιγότερο θανατηφόρα λόγω του συστήματος προειδοποίηση που λειτουργήσε χάνει στην προετοιμασία τη ε, κυβέρνηση και στον πληθυσμό που αντέδρασε σωστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Το κέντρο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής κινητοποιήθηκε αμέσω. Ε, τρία εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για άμεση ενίσχυση και οι εμπειρογνώμονε τη Γενική διεύθυνση ΕΚΟ πήγαν επί τόπου για να αξιολογήσουν τις ανάγκες. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαρίσω την δημόσια άμεση αντίδραση της κυρίας Επιτρόπου Γεωργίευας που έφτασε χθες στο Σαντιάκο για επιτόπου επισκέψεις. Οι περισσότερες φυσικές ε, καταστροφές είναι ξαφνικά γεγονότα. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διατηρηθούν οι ζωές επιτόπου και να μειωθούν οι κίνδυνοι με μια καλύτερη Παρασκευή και προετοιμασία και με ε, <clears throat> οικοδομές οι οποίες είναι ε, προγραμματισμένες για να αντέξουν αυτές τις ε, καταστροφές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουλίστα Ελκίζα. Εξ των ε, Δημοκρατών για τρία λεπτά. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχώς ε, εξ ονόματος της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής στην αλληλεγγύη μας για το λαό, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Χιλής για την καταστροφή την οποία υπέστησαν μετά το σεισμό και, και τα θύματα. Σου, τουλάχιστον 500 ε, θύματα χάθηκαν, αρκετοί Ευρωπαίοι μεταξύ αυτών και πάρα πολλές χιλιάδες τραυματίστηκαν. Τα χωριά Μαπούτσες ε, βρίσκονται σε ε, τρεις περιοχές της χώρας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν και όλοι τους επαγγελματίες που βοήθησαν τα θύματα. Οι αρχές της Χιλές στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων ενώπιον μιας τόσο δύσκολης κατάστασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την... Υπουργό Εξωτερικών της Χιλής, η οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα και να δράσει αμέσως ε, μετά από ένα σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε σπίτια και ε, ε, μας έδωσε τόσα θύματα. Και μαζί με την κυβέρνηση, η οποία έδρασε αμέσως, είχαμε και την αλληλεγγύη και της... Ε, ε, και των στρατηγικών τους εταίρου και με τους γείτονέ τους. Να ε, συγχαρώ και τη νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Πινέρα που σήμερα αναλαμβάνει καθήκοντα και να πω ότι θα πρέπει να του δώσουμε όλη τη στήριξη που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Χιλή είναι μια χώρα φίλο και είναι και μια χώρα η οποία ε, ανήκει στον ΟΣΑ θα φτάσει το ύψος της βοήθειας στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Επομένως ε, ζητώ να δοθούν στη διάθεση των αρχών της Χιλής όλα τα μέσα που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσει να ανοικοδομηθεί. Χρειαζόμαστε διεθνείς πιστώσεις ε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με το οποίο μόλις υπέγραψε συμφωνία η Χιλή θα πρέπει να συνδράμει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας Συγγνώμη, διακόρτει ο Πρόεδρος. Μήπως θα μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας ε, σύστησε ένα μηχανισμό ε, και ένα πυρήνα μετά του σεισμού, αντιμετώπιση των σεισμών και θα μεταβεί και η αρμόδια επίτροπος για να δει τι γίνεται επίτόπου στις επόμενες μέρες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και άλλες πολύ σημαντικέ δεσμεύσει όπως την ΑΕΤ βέβαια, αλλά θα πρέπει να σταθούμε και στο ύψο των περιστάσεων ε, μετά από όσα συνέβησαν στη Χιλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίγα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αλληλεγγύη προς μια χώρα μετά από μια καταστροφή όπως ε, αυτή την οποία συνέβησε στη Χιλή ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να δίνουμε οπωσδήποτε. Η Χιλή για μας ήταν μια χώρα η οποία μας υποδέχθηκε και προσέφερε άσυλο. Εκεί ζει μια μεγάλη κοινότητα Βάσκων που χρειάστηκε να μετικήσει στο 19ο αιώνα για οικονομικούς λόγους και στον 20ο αιώνα για πολιτικούς λόγους. Επομένως τα λόγια σε αυτέ τι περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από πράξεις. Και Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε αμέσως, απέστειλε 3 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση δράσεων και επίσης θα ήθελα να συγχαρώ και την αντίδραση της είπα της εκπροσώπου, της κυρίας Άστον, καθώς επίσης και της Επιτρόπου, η οποία έδρασε αμέσως και ήδη από χθε ε, είναι επιτόπου και εμψυχώνει και βλέπει τι ανάγκες υπάρχουν επιτόπου. Χαίρομαι επίσης και για τη λειτουργία του νέου συστήματος προστασία της ΕΚΟ, την ε, ε, βοήθεια που μπορέσαμε να δώσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και μέσω των διαφόρων οργανισμών μας. Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να παγιώσει το ρόλο της ως ε, δρα... Ε, συγκεκριμένος παράγων ε, στα θέματα αυτά συνεργαζόμενοι άμεσα με τους πληχθέντες και επίσης με τις διάφορες περιοχές. Θα ήθελα να ε, τονίσω τη δράση της Προέδρου Μπασιλέρη, η οποία για άλλη μια φορά απέδειξε πώς πρέπει να γίνεται η πολιτική. Θα πρέπει να δίνουμε, δείχνουμε ταυτόχρονα ανθρωπιά και φαντάζομαι ότι αυτό θα το μεταλαμπαδεύσει και στο νέο Πρόεδρο, στον κύριο Πινιέρα, που ελπίζω ότι θα δώσει και αυτό την ίδια όθηση για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η χώρα. Θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να εκφράσω την αλληλεγγύη μου, την υποστήριξή μου Προς όλα όσα έγιναν, προ όλε τι δράσει, ε, τα συλληπιτήριά μου στι οικογένειε των 500 θανόντων και ε, την αλληλεγγύη μου προ όλου όσους έμειναν άστεγοι. Η μία αντιπροσωπεία της ε, ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής μετέβη επιτόπου πριν από το σεισμό και είδαμε ότι είναι μια αντιπροσωπεια της ομάδα Ευρωπαϊκή Ένωση χιλης μετεβη επιτοπου πριν απο το σεισμο και ειδαμε οτι ειναι μια χωρα η οποία αποτελεί μοντέλο πρότυπο για την ανάπτυξη και ελπίζουμε ο σεισμός αυτός να μην ανακόψει αυτή την πορεία της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω προσυπογράφοντας ε, τα όσα είπαν οι συνάδελφοι Μουνής και Βουλπάου, διότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς την ε, ε, Χιλή και προς την κυβέρνηση της Χιλής, που πολύ σωστά εκπροσωπούν η πρόεδρος Βασιλέρ και ο νέος πρόεδρος αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ε, το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές δεν κάνουν διακρίσεις και δεν γνωρίζουν ποιος είναι πλούσιος ή φτωχός. Καταδικάζουν ανεξαιρέτως. Και φυσικά βέβαια οι φτωχοί πλήττονται ακόμα περισσότερο και είναι ε, απαραίτητο λοιπόν να γίνουν πολύ περισσότερα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν ε, τα απαραίτητα προστοζήν. Το τι θα κάνουμε μετά από την καταστροφή ε, δεν είναι το μόνο που πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν και ορισμένα διαρθρωτικά στοιχεία και εδώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση κύριε Επίτροπε. Με ενδιαφέρει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα Έχουμε ένα έγγραφο με τη Χιλή, προβλέπονται 40 εκατομμύρια ευρώ για τα χρόνια από το 2007 το 2013 και θα ήθελα να ξέρω ποια κονδύλια από αυτά θα διατεθούν για να ενισχύσουν τις δομές, ε, κυρίως σε θέματα υποδομών, ε, ε, αυτοκινητοδρόμους κτλ. Ποια κονδύλια θα δοθούν για την ανοικοδόμηση των κατοικιών, ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά τα τέτοια φαινόμενα να είναι πιο κατάλληλα προετοιμασμένη η χιλή για να τα αντιμετωπίσει. Και επίσης ποιοι από αυτούς τους πόρους έχουν ήδη διατοθεί προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο σεισμός κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και κατέστησε άλλους άστεγους. Θέλουμε να εκφράσουμε την ελληνική μας προς τη χώρα αυτή και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί ακόμη δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και άλλα βασικά αγαθά. Επίσης έχουν σημειωθεί καταλυστεύσεις και σε σπίτια και σε μαγαζιά. Πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε την αναγκή μας προς το λαό της Χιλής και να διασφαλίσουμε ότι οι ληστές θα τιμωρηθούν χωρίς να ξεχνάμε ότι στη χώρα αυτήν υπάρχουν τόσο απομακρυσμένες περιοχές που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί οι ανθρωπιστικές αποστολές. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη βοήθεια από την Ένωση, πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί χορήγησης βοηθείας για όλους όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Είναι πολύ ωραίο ότι μπορούμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη, αλλά να μην μείνει αυτό στα λόγια και να η στήριξη να υπάρχει και για το μέλλον. Ο κύριος Προβέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή ανάρρωση σας εύχομαι. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλους όσους πλήχθηκαν από αυτή την ε, φυσική καταστροφή. Δυστυχώς οι τραγωδίες ε, συνεχίζονται με αυτούς τους σεισμούς ε, πολλών ρίχτερ. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε θέματα κτηρίων και υποδομών. Έχουμε πάρα πολλού νεκρούς και επομένω αυτό που είναι σημαντικό είναι να συντονίζονται όλο και περισσότερο οι δυνάμει πολιτικής προστασίας για να μην ε, ε, υπάρχουν απώλεια πόρων και δεν, ε, να μπορούμε να δράσουμε αμέσω η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε πολύ γρήγορα στη Χιλή, αλλά θα πρέπει να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να μπορέσουν να συντονιστούν οι, εργασίες τους πάρα πολύ καλά. Σήμερα έφτασε στον τύπο η ειδησή ότι η το 50% της βοήθειας που δόθηκε στη Σουμαλία... ε, καταλυστεύτηκε από Ισλαμικές δυνάμεις, από τοπικές αρχές. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συλλογή ε, δημοσίων και ιδιωτικών δωρεών και επίσης την κατανομή της βοήθειας ε, στον πληθυσμό. Η γενεοδορία δεν θα πρέπει να προδίδεται και θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα υποπτίες προκειμένου να μην υπάρχουν ε, καταλυστεύσεις και να μην ξεχνάμε ότι ορισμένες φορές η βοήθεια φτάνει σε πολύ μακρινέ χώρε και μπορεί να αποδυναμωθούν οι δομές αυτές λόγω της κρίσεως. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντότς για δύο λεπτά. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα χαρούν όλοι να ακούσουν ότι υπήρχε θετική δράση στη βοήθεια προς τους ε, ανθρώπους εκεί στην Χιλή. Όλοι συγκινηθήκαμε από το πρόβλημά τους, αλλά θα ήθελα εγώ να στραφώ σε πιο γενικά θέματα που αφορούν γενικά την ανθρωπιστική μας στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περήφανη που είναι μέσα από τους δωρητές για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, θέλει να διασώσει ζωές, ε, να προσπαθήσει να φροντίσει να είναι όλοι έτοιμοι για την ανεπτώπιση φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά είναι πολύ καλέ προσδοκίε. Αλλά τα χρήματα που δίνονται δεν είναι τη Κομισιόν, είναι βρετανικά, γερμανικά, γαλλικά, από 27 δηλαδή χώρε. Σε μια εποχή οικονομική κρίση. κάθε μία από αυτέ τι χώρε θα πρέπει να αναγνωριστούν για τι προσπάθειε του. σω τα έγγραφά τη η Κομισιόν θα πρέπει να το αντικατοπτρίζει και να αναγνωρίσει τι προσπάθειε εκείνων που κάνουν, τα βάλουν αυτέ τι προσπάθειε δεν είναι η πολιτική και η ηγεσία του στον περλεμό που πληρώνουν, αλλά ο κάθε πολίτης, ο κοινός άνθρωπος. Ε, είναι αληθές ότι χρειάζονται ε, οι χώρες αυτές επίσης την ενίσχυσή μας για τη δημιουργία και διατήρηση δημοκρατικών δομών, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζονται επίσης την, την ε, βοήθειά μας για να τονίζουμε τα σφάλματα πολιτικών καθεστώτων που ε, οδηγούν στο ότι οι πολίτες ζουν πάντα σε ένδια στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόσφατος καταστροφικός και τόσο μεγάλης έντασης σεισμός στη Χιλή, πολύ λίγο χρόνο μετά από την καταστροφή στην Αϊτή, στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδε συνανθρώπου μα και επέφερε σημαντικό πλήγμα στι δομέ τη χώρα ιδίω στην περιοχή κονσεψιόν. οφείλουμε να σταθούμε δίπλα και στεκόμαστε στου πληγέντε και τι οικογένειέ του απερίφραστα δηλώνουμε την αλληλεγγύη μα. οφείλουμε να σταθούμε κοντά σε μια χώρα που μα συνδέουν στενοί φιλικοί δεσμοί και που αποτελεί μια από τι ισχυρότερε οικονομίε τη περιοχή πρότυπο ανάπτυξη για τι γειτονικέ χώρε αυτό το έχουμε διαπιστώσει και στα πλαίσια τη μεικτή διακοινοβουλευτική επιτροπή. θυμίζω ότι η ευρωπαϊκή ένωση και η χιλή έχουν υπογράψει συμφωνία σύνδεση η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2005 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η πολιτική και οικονομική συνεργασία αλλά και από κοινού ανάληψη δράσεων σε παγκόσμια κλίμακα εξάλλου η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει θεσπίσει ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τη χιλία αναφέρθηκε ήδη με εξαετή διάρκεια από το 2007 μέχρι το 2013 στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα απορρόφησης κοινοτικών πόρων από τη χώρα της λατινικής αμερικής για περιφερειακά για θεματικά προγράμματα που αναλαμβάνει η κυβέρνηση της χώρας η οποία μόλις πρόσφατα εξελέγη. η άμεση ανακοίνωση χρηματικής υποστήριξης και όλα όσα άλλα αναφέρθηκαν σήμερα από την επιτροπή μα. Ε, είναι ενθαρρυντικά θέλω όμως να τονίσω ότι για την ταχύτατη αντιμετώπιση και των συνεπειών αυτού του πρόσφατου σεισμού στις υποδομές της χώρας αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας οφείλουμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε την αποδέσμευση των προβλεπόμενων ε, πόρων και από το προαναφερόμενο στρατηγικό πλαίσιο ε, ευρωπαϊκής ένωσης χιλής. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς το λαό της Χιλής. Μια αλληλεγγύη την οποία εκφράσαμε και προς το λαό της Αιτής, της Τουρκίας και του Περού που πλήχθησαν από πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Η αλληλεγγύη καταδεικνύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα πρέπει να την διατηρήσουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα και στο μέλλον. Η Χιλή είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανταπόκρισης ε, σε φυσικές καταστροφές, αλλά ε, αυτές τις δυνατότητες δεν τις διαθέτουν οι περισσότερες περιοχές του κόσμου. Γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Η απάντησή μας μπορεί να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, πολύ πιο γρήγορη και πιο ε, αποδοτική εάν οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ποια είναι αυτή η κατεύθυνση. Κατ' εμέ θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών στις ε, διάφορες ε, υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Τρίτον, μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών και ανθρωπιστικών δράσεων. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ασφάλεια των ε, πολιτών και την, να τους δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρείται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της ανθρωπιστικής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο. Και τέλος, στα καθημάς, εάν θέλουμε η ανθρωπιστική βοήθεια και η απάντηση στην κρίση να αποτελεί σημαντικό άξονα της ανταπόκρισής μας, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, τόσο οικονομικούς όσο και ανθρώπινους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση Μπαρνιέ και να δημιουργήσουμε ένα ταμείο εθελοντισμού σε Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή είναι εδώ ο Επίτροπος ε, θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να συνδέσουμε περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια και την βοήθεια που γίνεται για ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χίγκιν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο, ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Στην αρχή σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγούσε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Μα 3 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής. Ευτυχώς ακούσαμε και άλλα. Το πρωί σήμερα ακούσαμε όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του σεισμού στη Χιλή και τους μετασυσμούς. Ξέρουμε ποια είναι λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία και ποιες είναι οι ανάγκες. 500.000 σπίτια έχουν καταστραφεί που πρέπει να ξαναφτιαχτούν. Ξέρουμε ότι ο ποιος είναι ο αριθμός των νεκρών και των αστέγων και εδώ μιλάμε λοιπόν για γενικό λογαριασμό 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και άρα η εισφορά μας πρέπει να είναι πολύ ψηλότερη από την αρχική. Στη συνθήκη της Λισαβόνας και ξέρετε ότι η Ιρλανδία είχε απορρίψει την πρώτη της μορφή πρέπει να προβλέπονται πολύ πιο συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης και γρήγορης αντιμετώπισης τέτοιων θεομηνιών αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς μεταξύ λόγων και έργων. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και να επανέλθει η ηλεκτρική ενέργεια και τα σπίτια τους να ξαναφτιαχτούν. Ευχαριστώ. Τώρα η οφθαλμοθυρία, ο κύριος Ρομέρα νομίζω ότι είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εχθές μίλησα με τον γερουσιαστή Χόρθε Πιθάρο, ο οποίος εδώ και κάποιες ώρες είναι πρόεδρος της Γερουσίας της Χιλής. Ο Πιθάρο σήμερα θα παραδώσει την ε, ε, προεδρική σκητάλη στον κύριο Πινέιρα και ελπίζω ότι θα κάνουν τα πάντα για την ανοικοδόμηση. Να συγχαρώ και την Πρόεδρο Βασιλέρ για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και την αδελφική μου στοργή προς το λαό της Χιλής για τις ε, πάρα πολύ σκληρές θεομηνίες, τους σεισμούς, ε, τα τσουνέμι, τα οποία χτύπησαν στην Κοθεπιόν, στο Βιομπίο και στο Βαλπαραΐσο. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι ο ερωικός λαός της Χιλής θα μπορέσει να ξεπεράσει όπως και άλλες φορές αυτή τη δραματική κατάσταση. Επαναλαμβάνω τη στοργή μου, την αγάπη μου και τη μεγάλη μου αλληλεγγύη. Thank you. Herr bitte. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταστροφικές συνέπειες ε, του σεισμού του 8,8 Ρίχτερ, θα πρέπει να ε, κατηγορήσουμε εκείνου που έδρασαν εκεί στην Κωνσηψιόν κατόπιν, γιατί 24 ώρες να περιμένει κανένας ε, μέσα στα ερήπια είναι πάρα πολύ χρόνος. Η βοήθεια έφτασε λόγω προβλημάτων λογιστικής ε, και οργάνωσης πάρα πολύ αργά. Και οι ομάδες που έφτασαν εκεί για βοήθεια δεν μπορούσαν να πέσουν το χάος, και οι πολίτες εκεί αναγκάστηκαν να διαφύγουν στις σκεπές των σπιτιών τους γιατί φοβόντουσαν τις πύρες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους ασίδωτες. Πρέπει να τους βοηθήσουμε εκεί, ναι, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε μία επίγουσα ανάγκη εξαφανίζεται η χρειά του πολιτισμού και βρισκόμαστε γυμνοί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και την πραγματικότητά μα. Θα πρέπει στο μέλλον η βοήθεια τη ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. So now I would like to ask... Ευχαριστώ κύριε Μόλτσερ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ποτότσνικ για να απαντήσει σε κάποιες παρατήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε βουλευτέ, σα ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή όλους μας όκορε το εύρος της ανθρώπινης αυτής καταστροφής με την ανταπόκριση από το ΕΚΟ μπορέσαμε να συντονίσουμε την πρακτική βοήθεια επιτόπου λίγο μετά από το πλήγμα του σεισμού. Η βοήθεια που δόθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διάφορα κρατημέλη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκτό από τι ανθρωπιστικέ και άλλε δράσει που προανέφερα, θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Χιλή, αναφέρθηκε αυτό, υπέγραψαν μια συμφωνία για να μπορέσει η τράπεζα αυτή να δρά και στην Χιλή. Αυτό αποδεικνύει τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής και οι προσπάθειες να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε την εταιρική μας αυτή σχέση. Είναι και πάρα πολύ ευκταίο γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό μέτσο που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει στην ανοικοδόμηση της χιλής. Όσον αφορά τη στρατηγική για την χιλή και τα χρήματα που δίνονται, έχω να πω ότι 25 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην πρώτη ε, στην πρώτη δόση και 15,6 παραμένουν για τη δεύτερη και θα μοιραστεί αυτό 50% για την οικονομική, της κοινωνικής συγγνώμη συνοχή και το άλλο 50% για την οικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως χρειαστούν τελικά για την ανοικοδόμηση. Η χιλιανή κυβέρνηση δεν ζήτησε συγκεκριμένη βοήθεια ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανοικοδόμηση. Ο πρόεδρος κ. Παίρνει αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του. Θα πρέπει να έχει το χρόνο να αξιολογήσει, να ποσοτικοποιήσει το, τις καταστροφές και να δει ποιες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να εξετάσει οποιοδήποτε αίτημα ε, ενδεχομένω υποβληθεί. Όπω ανέφερα προηγουμένω, το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσει τώρα να δράσει στην Χιλή μα δίνει ένα συμπληρωματικό μέσο για να βοηθήσουμε από εκείνο που είχαμε μέχρι στιγμή. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια, ένα καλό παράδειγμα η Χιλή, ο Υπουργός ε, Οικονομικών που αποχώρησε την ε, περασμένη Παρασκευή, τόνισε ότι εν αντιθέσει προς άλλες καταστροφές που έπληξαν τους ε, χιλιανούς, αυτή τη στιγμή οι χιλιανοί έχουν τους δικούς τους πόρους. Εν κατακλείδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες, οι περιφέρειες και οι χώρες της Ένωσης βρίσκονται ενωμένε με τη χιλή για να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή. Και έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα σε ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση εδώ, συνάδελφοι. Διακόπτει η συνεδρίαση μέχρι τις ψηφοφορίες στις 12 το μεσημέρι ακριβώς.